Ladies and gentlemen, let us start. Να αρχίσουμε κυρίες και κύριοι. Good morning to everybody. Καλημέρα σε όλους σας. Thank uh, Πρόεδρος, πριν, αρχίσω τις αποφ... πριν ε, διαβάσω τις αποφάσεις των συντονιστών, να σας υπενθυμίσω ότι θα χρειαστείτε σήμερα τις ε, ε, κάρτες της ψηφοφορίας σας, γιατί έχουμε ψηφοφορίες μπροστά μας. Να σας πω λοιπόν ότι μετά από αίτημα του εισηγητού το σημείο 15 θα μετατεθεί. έτσι ώστε να ψηφίσουμε, έτσι ώστε να ψηφίσουμε σε μία εβδομάδα για τις μικρές προσφυγές. Ε, αποφάσεις των συντονιστών τώρα. Η εισηγήτρια για τα, των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, θα ε, έρθει εδώ στις 15-16 Μαΐου, μάλλον όχι, θα την ακούσουμε μέσω video conference το ζήτημα των αποστολών και των ακροάσεων για το έτος 2015. Το πρόγραμμα θα σας το στείλουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ε, ο εισηγητής για τον προϋπολογισμό του 16 θα είναι ο πρόεδρός σας. Μια έκτακτη συνεδρίαση ενδεχομένως θα ε, γίνει στις 27 Απριλίου το απόγευμα. Θα κληθεί η Λουξεμβουργενή Προεδρία στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας το μήνα Ιούλιο. Η νομική υπηρεσία θα κληθεί να μας κάνει μία παρουσίαση όσον αφορά το νομοθετικό screening. Εκπρόσωποι των της ε, Επιτροπής μας ε, για, τα, ε, για την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για Ανθρώπους με Αναπηρία θα είναι η κυρία Χαουτάλα. Άλλο θέμα, ανεπίσημη συνεδρίαση με την Κομισιόν και το ΔΕΚ θα γίνει μετά από την συνάντηση των Σχιωδών την 27η Απριλίου στο Στρασβούργο. Όσον αφορά τις γνωμοδοτήσεις, η κυρία Χαουτάλα αναλαμβάνει την γνωμοδότηση για την προστασία κατά της εξωχωρικής εφαρμογής της νομοθεσίας που έχει ε, αναλυθεί από τρίτες χώρες και ο κύριος Ντουντά θα αναλάβει την γνωμοδότηση προς ε, ε, μία πράξη συνδεδεμένης ενιαίας αγοράς. Αυτές είναι οι αποφάσεις των συντονιστών και επομένως τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 14, σημείο 14 της σημερισίας διατάξεως, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την νομική προστασία κτλ. έχετε ε, όλοι τις ε, κάρτες σας. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Όχι ακόμα. Ψηφίζετε. Οκ, okay, εντάξει. Πέρας της ψηφοφορίας. εγκρίθηκε. 21 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Το 15 είπαμε έχει μετατεθεί, σημείο 16. ενδυνάμωση κάποιων αρχών της ε, τεκμηρίου αθωότητας ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Sorry. We first, sorry, we first. Which is the Uh, sorry. Uh, so, amendment uh, number 65. Τροπολογία 65. Ε, διανατάσεως της χειρός ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 14 ψήφοι υπέρ, 9 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Τροπολογία Όχι, πάμε απευθεία στο συμβιβασμό 2, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα διανατάσεως της χειρός, υπέρ, κατά. Ε, νομίζω ότι και εδώ πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Επαλήθευση λοιπόν. I close the Adopted Εγκρίνεται 15 ψήφοι υπέρ, 8 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Προχωράμε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Το ίδιο αποτέλεσμα εγκρίνεται. Πάμε στο συμβιβασμό υπαριθμών 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Φαίνεται να εγκρίνεται και αυτό. Συμβιβασμός 4. Υπέρ. Κατά. αποχές σαφώς εγκρίνεται συμβιβασμός 4 ε, 5 συγγνώμη Α, όχι, όχι, λέει ο Πρόεδρος. Τροπολογία 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 83. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. αποχές απορρίπτεται. Δεκαοκτώ. Τροπολογία δεκαοκτώ. Υπέρ. Τροπολογία 18, έτσι είναι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 85, υπέρ. νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε. Η Ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Πέρασε. Και απερίφθη. 10 ψήφοι υπέρ, 12 ψήφοι κατά, 2 αποχές. Συμβιβασμός 8. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 92 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές Ε, θα ήθελα παρακαλώ να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Συμβιβασμός 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 15 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Ε, νομίζω ότι ασφαλές θα ήταν να κάνουμε μια επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και επομένως περνάμε στην τροπολογία 113, υπέρ, κατά. αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία της τροπολογίας 113. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 114. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Μάλλον εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να το τσεκάρουμε. Άρχεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 17. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβασμός 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 33, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, αλλά πριν από αυτό έχουμε τον συμβιβασμό 19. Ναι, συμβιβασμός 19, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Επίσης, ε, είμαστε 26 ψηφίζοντες. Mr. Buddha should not vote. Ο κύριος Μπούντας νομίζω ότι δεν πρέπει να ψηφίσει. Εγκρίνεται λοιπόν, λέει ο πρόεδρος. 37, yes? Yes, we just heard 37. Yeah. 39. 39. 39. 39. Πού είμαστε λέγαμε άστο, είναι τροπολογία 39, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, να το ελέγξουμε καλύτερα. Η ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν αρχίζεται η ψηφοφορία από τη τροπολογία 42 πέρας. Απερι... Τροπολογία 44 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 20 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. πέρας της πληροφορία και εγκρίνεται. Τροπολογία 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Α, είναι ε, ταυτόσημη. Όχι. Τροπολογία 5, 50 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση καλύτερα επί της τροπολογίας 59 Χρειαζόμαστε άλλη μία ψήφο, να ψηφίσουν όλοι. Και απερίφθη η τροπολογία αυτή. Τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η γνωμοδότηση στο σύνολό της ναι, η... ηλεκτρονική ψηφοφορία αυτή πρέπει να είναι άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία πέρας και εγκρίνεται Uh, uh, θα, συνεχίσουμε τώρα με το σημείο 17 άσκηση νομικού επαγγέλματος ε, στην Ισπανία διανατάσσεως της χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Σημείο 18 της ημερησίας διατάξεως. Η κυρία Χαουτάλα θέλει να πάρει το λόγο. Ναι, παρακαλώ. Ήθελα να πω ότι κατά την άποψή μου δεν υπάρχει κανένας λόγος ε, να ε, αντιταχθούμε στη νομική βάση έτσι όπως αυτή έχει προταθεί. Ωστόσο θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θα πρέπει να συστήσει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να μην τροποποιηθεί η νομική βάση έτσι όπως έχει προταθεί από την Κομισιόν ε, παρά μονάχα σε περίπτωση που ε, τροποποιηθούν τα στοιχεία τα οποία περιέχονται στην πρόταση. Ε, συμφωνώ λοιπόν όσον αφορά την νομική βάση, αλλά λέω ότι ενδεχομένως εάν υπάρξουν στο μέλλον αλλαγές από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τότε ίσως θα πρέπει να συμφωνήσουμε και με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις που έχει προτείνει η Επιτροπή Περιβάλλον. Ο κύριος Φως. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι η απόφαση τώρα είναι καλή. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι και νομικά είναι λογικό. Όλες οι άλλες ενδεχόμενες σκέψεις θα ήταν υπόστατες Γι' αυτό επί της ουσίας βρίσκω ότι αυτή η τοποθέτηση είναι σωστή και γι' αυτό συμφωνώ. Πρόεδρος, εντάξει, θα ψηφίσουμε λοιπόν για να τάσω στους χειρός, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το σημείο 18 λοιπόν τελείωσε, το σημείο 19 όμως θα το ε, μελετήσουμε και κλεισμένο των θυρών. Επομένως όσοι δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε αυτή τη συνεδρίαση και κλεισμένο των θυρών παρακαλώ να εγκαταλείψουν την αίθουσα.